Σήμερα, συνάδελφοι, και αντικαθιστώ τον πρόεδρό μα, ο οποίο δυστυχώ δεν μπορεί να το. Το πρώτο θέμα, λοιπόν, που έχουμε στην ημερήσια διατάξη από χτες, έχουμε την έκθεση για, για τις διαπραγματεύσει. διαπραγματεύσεις. Το πρώτο, λοιπόν, θέμα ήταν το ο τρίμερης διάλογος φυσικάλη. Η 23 Ιανουαρίου συζητήθηκαν τα πρώτα θέματα, προγραμματισμός, αναφορές, αξιολόγηση, συνεργασία με τις λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνια και συνεργασία εξωτερικών εμπρεγνώμων, προγράμματα, δράσεις, εφαρμογή σε ό,τι αφορά τις ε, κατεξουσιοδότησης πράξης. Ευρία εντολή δόθηκε για τη τεχνική εργασία και για τον επόμενο τριμερή διάλογο, ο οποίος ε, περιμένουμε να λάβει χώρα στις 21 Φεβρουαρίου. Ελπίζουμε να είναι Το επόμενο θέμα, η αναθεώρηση για τι επενδυτικέ εταιρείε. Ε, ο πρώτο διάλογο έλαβε χώρα για το πακέτο αυτό και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξήγησαν τις θέσει του για τα βασικά πολιτικά θέματα, συμπεριλαμβανομένου και το πεδίο εφαρμογή για το IF4 σε ό,τι αφορά του κανόνες ε, και σε ό,τι αφορά τα βασικά στοιχεία, σε ό,τι αφορά τις εταιρείε ε, τάξης 3 και τα θέματα ρευστοποίησης. Ε, δεν ε, ευρέθηκε συμφωνία για τα βασικά ζητήματα. Το Κοινοβούλιο όμως και το Συμβούλιο εξέτασαν ενδεχόμενε πιθανότητε συμφωνήσει και ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί προ την κατεύθυνση αυτή. Συμφωνήθηκε να διατηρηθεί η συνοχή με τις πρόσφατα επιτευχθήσεις συμφωνίες για τα άλλα ζητήματα για τις τράπεζες. Επόμενος τριμερής διάλογος, αρχέ Φεβρουαρίου. Τρίτο θέμα, η συζήτηση για τριμερής διάλογος για τις εταιρικές, ε, τα εταιρικά ομόλογα. 23 Φεβρουαρίου, 21 Φεβρουαρίου θα λάβει χώρα για τις διατάξεις ε, σε ό,τι αφορά τα παράγωγα κτλ. Συζητήθηκαν όλα αυτά εκτενώς και Επίσης συζητήθηκαν τα μεταβατικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τον κανονισμό, σε ό,τι αφορά και τις ε, πατερικά ομόλογα. Είναι η πρώτη φορά όμως που συζητήθηκε το θέμα αυτό. Προγραμματίζονται περίπτερα τρίμερες διάλογοι για τον Φεβρουάριο. Αυτά λοιπόν στο σημείο 3, το οποίο αναβλήθηκε από χτες. Ας ελέγξουμε λοιπόν για τις ψηφοφορίες. Να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Δεν έχει ο κύριος Λούκα την κάρτα. Θα το λάβουμε υπόψη. Μάλιστα. Τρεις ψηφοφορίες. Πρώτη. Οι υποχρεώσεις ε, ευστοποίησης ό,τι αφορά του κύριου Γκολτιέρη. Το πρώτο λοιπόν θέμα. Παραγραφός 1 και 2 έχουμε το πρώτο θέμα. Υπέρ. Κατά. Συμφωνείτε, εγκρίνεται. Ετρολογική σκέψη 9 ως 9 μπορούμε να ψηφίσουμε με μπλοκ. Υπέρ. συμφωνείτε, κατά. Εγκρίνεται. λογικέ σκέψει α, β και γ. Μαζί τα ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Και ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιηθήκε. Με ονομαστική κλίση. Ζητώ συγγνώμη. Including Mr. Luca. Και ο κύριος Λούκα. Πέρασε. Πολύ ωραία. Εγκρίνεται με σημαντική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Γκουαλτιέρη. Δεύτερο θέμα. Συμβάσεις παραγόγων OTC που δεν έχουν περάσει από το IPC, παράγραφος 1 και 2, μαζί ψηφίζουμε παρακαλώ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 1 έως 12, τηλεγικές σκέψεις, αν μπλοκ παρακαλώ ψηφίζουμε υπέρ, κατά εγκρίνεται. Και α, β και γ, αμπλόκ υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Και το κείμενο όπως τροποποιήθηκε τώρα με ονομαστική κλίση. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. 35 ψήφοι υπέρ, μία κατά 6 εποχές. Ευχαριστώ. Και τελική ψηφοφορία. Άλλη μία στάση για τις ε, υποχρεώσεις που σχετίζονται με τον Brexit. Παράγραφος 1 και 2 unblock ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 9 έως 10 αιτιολογικές σκέψεις unblock υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και αιτιολογικές σκέψεις α, β, γ υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Το κείμενο αποστροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρα ψηφοφορίας. 35 ψήφοι υπέρ. 7 αποχές, καμία κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Σα ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Επόμενη συνεδρίαση στι 4 Φεβρουαρίου, Δευτέρα, από 3 μέχρι 6.30 υπό επιβεβαίωση όμω.